D'après. Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Möchte nicht in die Tag. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αρχίζει η συνεδρίαση. Δεν θέλω να μπούμε στην ημερήσια διάταξη. χωρίς να εκφράσουμε κι εμείς ε, τον αποτροπιασμό μας για την ε, βιότητα με την οποία δολοφονήθηκε χθε ε, ένας στρατιώτης της ΗΠΑ και θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο να μεταφέρει την, τα συλληπιτήριά μας, τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Δεν συνηθίζεται να παίρνω το λόγο, αλλά έχω ένα ερώτημα που πρέπει να θέσω στους φίλους σοσιαλιστές. Έχει τελειώσει στη Βουλγαρία η προεκλογή.